ο λόγος των εκπρόσωπο του Συμβουλίου. Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, την Παρασκευή 26 Ιουνίου, μια μαύρη μέρα της ιστορίας ε, που σημαδεύτηκε από πολλαπλές τρομοκρατικές επιθέσεις, ε, τρεις ε, χώρες χτυπήθηκαν σχεδόν ταυτόχρονα η Γαλλία, το Κουβέιτ και η Τινησία. Αυτές οι τρομοκρατικές επιθέσεις μία ακόμα φορά μας υπενθύμησαν ε, τον βρώμικο χαρακτήρα της τρομοκρατίας ε, και κυρίως ε, αυτών που εκτελούν τις τρομοκρατικές πράξεις τις διατάζουν. Η αντίδρασή μας θα πρέπει να είναι αλληλέγγυα και αυστηρή. Ε, Στι 26 Ιουνίου ήδη το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο είπε ότι θα πρέπει να ενισχύσουμε τη δράση μας ε, ενάντια σε αυτές τις τρομοκρατικές απειλές. Αυτός ο αγώνας εναντίον της τρομοκρατίας αποτελεί για τις ανοιχτές μας και δημοκρατικές μας κοινωνίες μία από τις πιο σημαντικές προκλήσεις για το μέλλον. Συνεπώς, μία από τις πρώτες μας προτεραιότητες ε, της Προεδρία μα, τη Προεδρίας του Λουξεμβούργου, είναι αυτή ακριβώ και θα βασιστούμε στι εργασίε των προκατόχων μας, λαμβάνοντας ε, υπόψη τόσο τι εσωτερικέ όσο και τι εξωτερικέ πτυχέ της ασφάλεια. Η Λουξεμβουριανή Προεδρία θα προσπαθήσει έτσι ώστε η Ευρωπαϊκή Ένωση να υιοθετήσει μια συνεκτική προσέγγιση στην καταπολέμηση τρομοκρατίας ε, που θα περιλαμβάνει και τις εσωτερικές και τις εξωτερικές πτυχές της ασφάλειας. Ε, συνεργασία η οποία θα πρέπει να λάβει χώρα μεταξύ των κρατών μελών, της Κομισιόν, την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης ε, και τον συντονιστή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Διαθέτουμε εργάνω όπως η Europol, η Eurojust, η Frontex ε, και η SEPOL. Θα πρέπει να δώσουμε σε αυτά τα όργανα, σε αυτούς τους φορείς, τα μέσα και τους πόρους που είναι απαραίτητοι. Ω απάντηση στι τρομοκρατικέ επιθέσει του, του Παρισιού τον Ιανουάριο, οι αρχή κρατών κυβερνήσεων στι 12 Φεβρουαρίου υιοθέτησαν μια δήλωση που βασίστηκε σε τρει πυλώνε. Να διασφαλιστεί η ασφάλεια των πολιτών, να προληφθεί ε, η, ε, ε, η ριζοσπαστικοποίηση ε, και η συνεργασία με τους εταίρους μας. Ε, το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο έλαβαν μια πλήρη έκθεση για την εφαρμογή αυτών των μέτρων από την, προηγούμενη, από την Κομισιόν. Στις 28 Απριλίου η Κομισιόν υιοθέτησε το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Ασφάλειας. Το συζητήσαμε μάλιστα χτες η καταπολέμηση της τρομοκρατίας είναι μία από τις ε, πρώτες προτεραιότητες. Η ισχυρή διεθνής διάσταση της τρομοκρατίας υπογραμμίστηκε και η δράση μας θα πρέπει να τοποθετηθεί ακριβώς στο ίδιο διεθνές επίπεδο. Αυτό σημαίνει ότι το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων ε, και γι' αυτό μάλλον το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων σε 9 Φεβρουαρίου υιοθέτησε συμπεράσματα για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας με στόχο να ενισχυθεί η συνεργασία με τις χώρες της Βόρειας Αφρικής, της Μέσης Ανατολής, του κόλπου καθώς επίσης και με την Τουρκία και τις χώρες των Βαλκανίων. Ένα αριθμός ε, σχεδίων ενίσχυσης των ε, δυνατοτήτων αντιμετώπισης τρομοκρατίας εγκρίθηκε. έγιναν και σεμινάρια στο Λίβανο και την Τουρκία ήδη για αυτό το θέμα ο συντονιστής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας ε, πήγε στην Τινησία επικεφαλής μιας διπηρεσιακής υπηρεσίας ε, κατόπιν ε, της οποίας η ανώτατη εκπρόσωπος ε, πρότεινε στον πρόεδρο της Τινησίας μια σειρά μέτρων. Επιπλέον, μια task force για την στρατηγική ενημέρωση δημιουργήθηκε και θα επεξεργαστεί μια στρατηγική επικοινωνίας προς τον αραβικό κόσμο. Πρέπει επίσης να συνεχίσουμε δραστηρία τη συνεργασία με τα Ηνωμένα Έθνη, το ΝΑΤΟ, το Συμβούλιο της Ευρώπης και άλλους διεθνείς οργανισμούς, καθώς επίσης και την διμερή συνεργασία με τους βασικούς εταίρους μας όπως οι Ηνωμένε Πολιτείες. Στις 16 Ιουνίου, οι Υπουργοί Εξωτερικών Υποθέσεων ε, συμπεράνουν ότι έχει επιτευχθεί σημαντική απτή πρόοδος ε, προκειμένου να προλάβουμε ε, της, ε, ε, την εξώθηση νέων ε, στις χώρες μας αλλά και σε γειτονικέ χώρες που, για την συμμετοχή τους σε τρομοκρατικές οργανώσεις. Εκεί πρέπει να δουλέψουμε σε βάθος και μάλιστα σε πολλά επίπεδα, στην εκπαίδευση, στην ενσωμάτωση, στις αρχές μας. Και γι' αυτό λόγο το κέντρο αριστείας θα, ένα κέντρο αιστείας θα δημιουργηθεί, αλλά θα ληφθούν και άλλα μέτρα, όπως για παράδειγμα ενίσχυση του πλαισίου της Σέγγεν, ε, σύμφωνα με το οποίο ε, έγγραφα και πρόσωπο και άτομα θα την χάνουν περισσότερο πιο ισχυρό ελέγχου με βάση μια προσέγγιση αξιολόγησης κινδύνου. Ήδη τον Ιούνιο ολοκληρώθηκε η προετοιμασία και θα εφαρμοστεί ήδη. Ε, μάλιστα ενημερώθηκαν και τα εγχειρίδια στα σημεία ελέγχου των συνόρων. Ε, επίσης παρακολουθεί το 1 Ιουλίου το περιεχόμενο στο ίντερνετ. Η Europol ε, παίδι να ενισχύσει την συνεργασία με τον, ε, ε, για, το, για το θέμα αυτό. Ε, θα πρέπει να παρακολουθούμε την ε, προπαγάνδα, εξτρεμιστική προπαγάνδα που γίνεται στο ίντερνετ και να την απαγορεύουμε, ε, σεβόμενοι όμως τα θεμελιώδη δικαιώματα. Το Συμβούλιο σύντομα θα υιοθετήσει μια απόφαση για την υπογραφή εκ μέρους Ευρωπαϊκής Ένωσης του προσθέτου πρωτοκόλου στην Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την πρόληψη της τρομοκρατίας που θα ε, ποινικοποιεί την χρησιμοποίηση ξένων ε, πολεμιστών. Ε, η συνεργασία με ε, τρίτες χώρες είναι επίσης πάρα πολύ σημαντική. Θα πρέπει να τις βοηθήσουμε να ε, καταπολεμήσουν και τις κοινωνικές αιτίες του, της τρομοκρατίας, όπως για παράδειγμα η ενέργεια των νέων, που δημιουργούν απελπισία στους νέους και τους καθιστούν έφοροι γη για τη στρατολόγηση τους από τρομοκρατικές ομάδες. Η Τινησία είναι δυστυχώς ένα τέτοιο παράδειγμα. Η Προεδρία του Λουξεμβούργου θα μεριμνήσει ε, και γι' αυτό το λόγο προτείνουμε την επόμενη εβδομάδα μια καινούργια πρωτοβουλία συνεργασίας με τις χώρες του Μαγκρέμπ για την, για την απασχόληση των νέων, για την κατάρτιση των νέων, διότι ε, θα πρέπει το πρόβλημα να το αντιμετωπίσουμε στη ρίζα του. Υπάρχουν νέοι οι οποίοι νιώθουν τον πειρασμό της τρομοκρατίας στη Συρία και αλλού εξαιτίας ε, της κατάστασης στην οποία βρίσκονται. Κυρίε και κύριοι, θα ήθελα να επανέλθω στο θέμα της ριζοσπαστικοποίησης. Ε, το φαινόμενο αυτό διαδίδεται και είναι ανησυχητικό. Μερικές ε, φορές οι νέοι ριζοσ, μέσα σε μια περίοδο δύο μηνών μόλις. Ε, θα, οργανώσουμε ένα συνέδριο για την επανένταξη και την ριζοσπαστικοποίηση παστικοποίηση στις φυλακές γιατί πολλές φορές από εκεί προέρχονται αυτοί οι νέοι τρομοκράτες. Ε, τι μεταχείριση θα πρέπει να επιφυλάσσουμε στους ξένους μαχητές που έρχονται στις κοινωνίες μας. Είναι ένα άλλο πρόβλημα που θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Η κυρία ε, Γεροβά, η Επίτροπος, ε, ε, τροποποίησε τη χρηματοδότηση έτσι ώστε η καταπολέμηση τρομοκρατίας να συμπεριληφθεί στον τομέα της δικαιοσύνης φέτος. Θα ενισχύσουμε τα μέσα για να ε, καταπολεμήσουμε τη χρήση του ίντερνετ και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης από τρομοκρατικές ομάδες ε, για να προωθούν την προπαγάνδα τους και για να στρατολογούν νέους. Θα στείλουμε μηνύματα αντίθετα με αυτή την προπαγάνδα και θα ξεκινήσουμε οργανωμένες εκστρατείες μέσα στο ίντερνετ και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Επίσης ε, θα ε, πρέπει να καταπολεμήσουμε τα πυροβόλα όπλα τη χρήση τους και να τα κατάσχουμε. Ε, θα πρέπει να αστούμε επίση στην ανταλλαγή πληροφοριών. Αύριο, στην άτυπο συνέδριο Υπουργών Δικαιοσύνη και Ιστορικών Υποθέσεων στο Λουξεμβούργο, θα αποφασίσουν για την βελτίωση τη ανταλλαγή πληροφοριών ανάμεσα στην αστυνομία και στι ε, υπηρεσίε πληροφοριών. Όπω σα είπα και χτε, ε, η εφαρμογή τη στρατηγική εσωτερική ασφάλεια ε, 15.020 ε, αποτελεί ε, προτεραιότητα της ε, εξωβρινής προεδρίας και μπορεί να γίνει πραγματικά χρήσιμο εργαλείο στην μάχη κατά της τρομοκρατίας. Θα πρέπει να είμαστε αποφασιστικοί και να αντιμετωπίσουμε καταρχήν τις βαθιές ρίζες του φαινομένου. Να μην πέσουμε στην παγίδα που μας στείλουν οι τρομοκράτες, δηλαδή να αποδυναμώσουμε τις αρχές μας και το δημοκρατικό μας σύστημα. Οι δημοκρατίες μας είναι, θα είναι πιο ισχυρές όταν η δράση μας σέβεται ε, τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ευχαριστώ πολύ. Ε, Ευχαριστούμε πολύ. Εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο κύριος Αβραμόπουλος έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αγαπητά μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, οι τρομοκρατικές ενέργειες της ε, Παρασκευής 26 Ιουνίου στη Γαλλία, την Ισία και Κουβέιτ, καθώς και στη Σομαλία, καταδεικνύουν για άλλη μία φορά τον απάνθρωπο χαρακτήρα των τρομοκρατών. Θα ήθελα καταρχήν εξ ονόματος της Επιτροπής να ε, εκφράσω τα συλληπιτήριά μου προς τις οικογένειες των θυμάτων και να εκφράσω την ε, ηθική μας υποστήριξη και τις, στις χώρες που έχουν πληγεί στην Ευρώπη και εκτός αυτής. Θα ήθελα να καταδικάσω αυτές ε, τις τρομοκρατικές πράξεις σε υψηλούς τόνους. Πρέπει να αντιμετωπίσουμε συλλογικά αυτή την απειλή. Θα πρέπει να προσδώσουμε ασφάλεια στους πολίτες μέσα στα πλαίσια των αξιών μας. Βεβαίως αντιμετωπίζουμε συνεχώς απειλές και τα πολυάριθμα θύματα των φετινών ε, τρομοκρατικών ενεργειών μας ε, ε, τονίζουν αυτή την πραγματικότητα διερενεργούνται ε, έρευνες από τις αρμόδιες εθνικές αρχές και από τις διαθέσιμες πληροφορίες μπορούμε να πούμε ότι οι, οι α, άνθρωπες αυτές τρομοκρατικές ενέργειες στη Γαλλία, την Ισία και Κουβέιτ δείχνουν μία απάνθρωπη ιδεολογία, μία ιδεχθή ιδεολογία μυσαλλοδοξίας Στόχος τους είναι να ενσταλλάξουν το, τον τρόμο. Οι τρομοκράτες έχουν σκοπό να πλήξουν ήπιους στόχους, δηλαδή ε, θρησκευτικά οικίματα ή ε, τουριστικά θέρετρα. Όπως ξέρετε, η Επιτροπή συνεργάζεται στενά με τα κράτη-μέλη για να ορίσουμε τομείς όπου η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί πραγματικά να αντιμετωπίσει την τρομοκρατία και τη ριζοσπαστικοποίηση. Αποτελεσματικά προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε αυτές τις απειλές. Τον Απρίλιο η Επιτροπή παρουσίασε την Ευρωπαϊκή Ατζέντα για την Ασφάλεια η ατζέντα έχει υψηλή, ως υψηλή προτεραιότητα την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας. Πρόκειται για μία έννοια ασφάλειας που περιλαμβάνει το κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα. Η ατζέντα αυτή ορίζει μία πληθώρα δράσεων για να αντιμετωπίσουμε την απειλή της τρομοκρατίας αρχίσαμε να εργαζόμαστε ε, ενεργά και δραστήρια για την ε, εφαρμογή τους. Θα ήθελα να σας ε, μιλήσω για την συνεχιζόμενη εργασία μας ύψης της πολιτικής και πρακτικής σημασίας. Η ριζοσπαστικοποίηση και αντιμετώπιση της είναι ύψης της σημασίας. Υπάρχει ένα κέντρο αριστείας μάλλον θα δημιουργηθεί το Σεπτέμβριο αυτό το κέντρο αριστείας για να αντιμετωπίσει το ζήτημα έμπρακτα. Θεωρώ ότι θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε την τρομοκρατία σε ευρωπαϊκό επίπεδο με βάση αντιτρομοκρατικές δυνάμεις. Επίσης, από την 1η Ιουλίου ε, ορίστηκε αυτό το λειτουργικό κέντρο της Europol που θα είναι ε, πλήρως λειτουργικό μέσα σε ένα χρόνο. Αυτό το κέντρο αναφοράς ε, θα ήθελε να αντιμετωπίσει τις αιστείες τρομοκρατίας έτσι ώστε να μπορούν να αρθούν οι κίνδυνοι. Μέχρι το τέλος του έτους η Επιτροπή επίσημα θα εκκινήσει μία ε, πλατφόρμα αντιμετώπισης της τρομοκρατίας μέσα στα πλαίσια του κυβερνοχώρου για να μειώσουμε την προσβασιμότητα, την επιγραμμική προσβασιμότητα του τρομοκρατικής προπαγάνδας στο διαδίκτυο και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Θα υπάρξει και ένα workshop στις 24 Ιουλίου με εμπειρογνώμονες από τη βιομηχανία και τις κοινότητες επικράτησης του δικαίου. Επίσης, η προστασία των εξωτερικών συνόρων είναι ύψης της σημασίας. Θα θέλαμε να βοηθήσουμε τα κράτη-μέλη να μπορέσουν να προωθήσουν αυτούς τους ε, ελέγχους μέσα στα πλαίσια μιας στοχοθέτησης έτσι ώστε να ορίσουμε ε, μία πρώτη σειρά δικτών κοινών κινδύνων. Η Europol και η Frontex θα ε, εφαρμόσουν αυτά τα δεδομένα και τώρα έχουμε αναθεωρήσει και το εγχειρίδιο για τους συνοριαφύλακες ως προς την, ε, το εγχειρίδιο αντιμετώπισης κινδύνων προωθούμε πληροφορίες και σε τελωνιακό επίπεδο, έτσι ώστε να ανοιχνεύσουμε τις ύποπτες διακινήσεις αγαθών. Πέμπτον, θέλουμε να ανοιχνεύσουμε τα δίκτυα χρηματοδότησης της ε, τρομοκρατίας και χρησιμοποιούμε και όλα τα κέντρα πληροφόρησης η πρόσφατη έγκριση της οδηγίας για την αντιμετώπιση των εσόδων από παράνομες δραστηριότητες έχει βοηθήσει προς αυτή την κατεύθυνση. Έκτον, όπως ορίζεται από την Ευρωπαϊκή Ατζέντα για την Ασφάλεια, θα πρέπει να προστατεύσουμε καλύτερα τους ε, πολίτες μας κατά των απειλών τρομοκρατίας. Αυτό σημαίνει ε, μια συγκεκριμένη εργαλειοθήκη καθώς και ε, ένα εγχειρίδιο κατευθυντηρίων γραμμών για την αντιμετώπιση αυτών των soft targets. Προσπαθούμε να αναθεωρήσουμε και να ε, προβάλλουμε αυτό το δίκτυο για την πρόληψη απειλών και ε, δίκτυα, μέσα από δίκτυα έγκαιρης προειδοποίησης και αντιμετώπισης. Έβδομο, Τη στιγμή που οι εναέριες κυκλοφορίες είναι αγαπητός στόχος των τρομοκρατών, προσπαθούμε να προωθήσουμε την ασφάλεια της ε, ε, εναέριας ε, κυκλοφορίας μέσα στα πλαίσια και των ζωνών σύραξης, ορίζοντας και συστάσεις προς τις αεροπορικές εταιρείες και το κοινό. 8 θα πρέπει να αναφέρω το Ευρωπαϊκό PNR που είναι αναπόσπαστο μέρος της ε, ατζέντα μας για την ασφάλεια. Θα ήθελα να ευχαριστήσω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τις προσπάθειες που έχει καταβάλει έτσι ώστε να ολοκληρωθεί η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία για το PNR για τα στοιχεία των επιβατών. Είμαι πεπισμένος ότι μπορούμε όλοι να συνεργαστούμε επικοδομητικά έτσι ώστε οι από κοινού νομοθέτες να αποφασίσουν επί ενός κειμένου υψηλής προστασίας δεδομένου, το οποίο θα είναι και αποτελεσματικό. Ένατον, οι πρόσφατες ε, τρομοκρατικές επιθέσεις ε, καταδεικνύουν ότι θα πρέπει να υπάρξει καλύτερη διεθνή συνεργασία και συντονισμός. Οι επιθέσεις στην Τινησία ε, ήταν συμβολικού χαρακτήρα διότι έπισε τον τουρισμό που είναι ένας τομέας ζωτικής σημασίας για τη χώρα. Επρόκειτο για μία επίθεση κατά της φιλοξενίας της Τινησίας και των μακροχρόνιων δεσμών της με την Ευρώπη. Θα πρέπει να υποστηρίξουμε τους Τινήσιους εταίρους και να δείξουμε αλληλεγγύη. Αυξάνοντας την ασφάλειά τους θα συνεισφέρουμε και στη δική μας. Υπό το φως των επιθέσεων στο Μουσείο του Μπαρτό συναντήθηκα στην Τίνιδα με τους ομολόγους μου για να δούμε πώς μπορούμε να υποστηρίξουμε ως Ευρωπαίοι εταίροι. Θα πρέπει να συνεργαστούμε για να ε, αντιμετωπίσουμε τις ρίζες της κακοδαιμονίας, της ρίζοσπαστικοποίησης, χτίζοντας ε, πλαίσια, ικανά πλαίσια αντιμετώπισης της τρομοκρατίας και των απειλών. Αγαπητά μέλη, έχουμε συνεργαστεί τους τελευταίους έξι μήνες και έχει επιτελεστεί πρόοδος σε πολλούς τομείς. Αλλά οι πρόσφατες τρομοκρατικές επιθέσεις μας υπενθυμίζουν ότι πρέπει να γίνουν ακόμα πολλά. Το χρωστάμε αυτό στα θύματα, στους πολίτες μας και στους εταίρους μας. Γι' αυτό ας συνεχίσουμε με αποφασιστικότητα να προβάλλουμε τις ε, κοινέ μας προσπάθειες για την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας και της ριζοσπαστικοποίησης. Ευχαριστώ. Ε, Ευχαριστώ πολύ κύριε Επίτροπε. Παίρναμε τώρα στους ομιλητές από τους ε, εκπροσώπους των πολιτικών ομάδων από το ΕΛΚ η κυρία Μόνικα Χολμάιερ έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ αγαπητοί συνάδελφοι. Τα πρόσφατα γεγονότα, οι τρομοκρατικές επιθέσεις μας έχουν δείξει ότι σε μια ανοιχτή και ελεύθερη κοινωνία μπορούμε να είμαστε ευάλωτοι. Κατέδειξε επίσης ότι, το, ότι στην άμεση γειτονιά μας, στη Μέση Ανατολή και στην Βόρεια Αφρική <clears throat> δεν υπήρχε ποτέ τόσο μεγάλη αναταραχή και τόσο βίαιες επιθέσεις όπως το παρελθόν. Γι' αυτό είναι απαραίτητο από τη μία πλευρά να συνεργαστούμε με τους εταίρους που είναι έτοιμοι να εργαστούν μαζί μας για να αντιμετωπιστεί η τρομοκρατική απειλή. Θα πρέπει να κάνουμε την προσπάθεια να προχωρήσουμε σε καλύτερη συνεργασία μαζί τους και γι' αυτό χαιρετίζω αυτά που ελέγχθησαν και από την Κομισιόν και από το Συμβούλιο. Είναι απαραίτητο λοιπόν να πάρουμε πολύ στα σοβαρά και πολύ οργανωμένα το πρόβλημα της ασφάλειας και επομένω να προχωρήσουμε στα κατάλληλα μέτρα. Ελπίζαμε να μην χρειάζεται να προσφύγουμε σε αυτά τα μέτρα, αλλά η σημερινή κατάσταση δείχνει ότι είναι απαραίτητο για να προστατεύσουμε τους πολίτες μας. Αυτό λοιπόν θα πρέπει να συνδυαστεί με το σύστημα PNR, με ένα νέο ευρωπαϊκό σύστημα το οποίο θα πρέπει να λειτουργήσει καλά ώστε να, μπορέσουν, να μπορέσει αυτό να καλύψει όλες τις ευρωπαϊκές χώρες και να συνεργάζεται με τρίτες χώρες ώστε έτσι να έχουμε μια καλύτερη εξασφάλιση των εξωτερικών μας συνόρων αλλά θα πρέπει εδώ να είμαστε και σαφείς ότι είναι δύσκολο να ανακαλύψουμε τους πράκτορες οι οποίοι βρίσκονται σε κατά κάποιο τρόπο ύπνωση ή βρίσκονται, έχουν διαβρώσει τις ε, μυστικές υπηρεσίες ή τα διάφορα τους άλλους φορείς της κοινωνίας και οι οποίοι είναι έτοιμοι να κινητοποιηθούν για να επιτεθούν κατά των πολιτών μας. Πρέπει λοιπόν να προσπαθήσουμε να βρούμε όλους αυτούς τους ανθρώπους και ιδίως να μπορέσουμε να σπάσουμε τα δίκτυα της ριζοσπαστικοποίησης στην Ευρώπη. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να αντιμετωπίσουμε τη ριζοσπαστικοποίηση και την ευκαιρία να χρησιμοποιηθούν τα άτομα για σκοπούς αντίθετους από τη θέλησή τους, όλα αυτά να τα αντιμετωπίσουμε με όλα τα μέσα τα οποία μας δίνει το κράτος δικαίου. Ευχαριστώ πολύ, λέω πρόεδρος, για την σοσιαλιστική ομάδα, η κυρία Τάνια Φαγιών. Έχετε το λόγο. Δύο λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Είναι σαφές ότι προφανώς πρέπει όλοι μας να καταδικάσουμε αυτές τις ενέργειες και θα πρέπει να ενώσουμε τις δυνάμεις μας για να μπορέσουμε να υποστηρίξουμε τις αξίες οι οποίες είναι σημαντικές για μας, όπως είναι η ισότητα, η ελευθερία, η ανεκτικότητα. Δεν είναι μονάχα το θέμα της ενίσχυσης τις ασφάλειες, αλλά πρέπει να αντιμετωπίσουμε και τα κοινωνικά προβλήματα που έχουμε ενώπιόν μας. Θα πρέπει να δούμε πού βρίσκονται οι ρίζες της τρομοκρατίας πρόκειται για την, στις χώρες αυτές. Είναι τα θέματα ένδυας, είναι τα θέματα των συγκρούσεων. Είναι λαθασμένο να πούμε ότι όλη η τρομοκρατία έχει θρησκευτικούς λόγους. Η τρομοκρατία ξεκινάει από την δυσπιστία, από τα στερεότυπα δεν γίνεται, δεν υπάρχει αγώνας μεταξύ της δύση και του Ισλάμ. Έχουμε Ευρωπαίους οι οποίοι πηγαίνουν στις χώρες αυτές στην, ε, στην Συρία και το Ιράκ αλλά εκεί πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι τα άτομα θα πρέπει να είναι πιο ενσωματωμένα στις κοινωνίες μας. Μόνο έτσι μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα αυτά. Το PNR μπορεί να είναι κάτι το οποίο χρειάζεται, αλλά δεν πρέπει να οδηγήσουμε σε μέτρα τα οποία αντιμετωπίζουν όλους τους επιβάτες των αεροπορικών εταιών σαν δυνητικούς ε, τρομοκράτες. Είμαι πεπισμένη λοιπόν αγαπητοί συνάδελφοι, Ο, είμαστε, υποχρεωμένοι να αγωνιστούμε κατά της ε, ε, τρομοκρατίας, αλλά αυτό τονίζοντας την αξία των ανθρωπίνων αξιών και της ελευθερίας έκφρασης και έτσι να ξεπεράσουμε το μίσος και το φόβο ο Τσάρλ Τάνοκ. ένα μισή λεπτό. Πρόεδρε, ε, την Ισία, Γαλλία, Κουβέιτ, διαφορετικά πράγματα, αλλά έχουν ένα κοινό παρανομαστή. Ε, όλοι οι τρομοκράτες ε, συνδέονται με τον ΆΙΣ, με τον Ισλαμικό στρατό. Ένα χρόνο μετά την αντιπίθεση του ε, ο χάρτης της Μέσης Ανατολής αλλάζει και μετά την απελευθέρωση του Κομπάνη, λίγο μετά την απελευθέρωση του Κομπάνη, το, Ισλαμικός ε, στρατός έκανε επιθέσεις και εκεί, τρομοκρατικές επιθέσεις, ε, θανατώνοντας ε, εκατοντάδες ανθρώπους πολλά, και πολλά παιδιά μεταξύ αυτών. Ε, η Συρία αποτελεί ένα καινούριο μαγνήτη τρομοκρατών. Ε, στο παρελθόν ξέραμε το μοντέλο της ε, Αλκάιντα ε, που βασιζόταν σε κάποια παράπονα που είχαν που παρόλο που δεν ήταν βάσιμα τώρα έχουμε το καινούργιο αυτό μοντέλο που οι τρομοκράτες επιτίθενται σε μειονότητες, σε άλλα θρησκεύματα περισσότερο από ό,τι σε συγκεκριμένα κράτη. Θα πρέπει να κάνουμε περισσότερα πράγματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση έτσι ώστε να διασφαλίσουμε ότι οι κοινωνίε μα θα είναι σε εγρήγορση και θα αντιμετωπίσουμε το θέμα τη στρατολόγηση. Θα πρέπει να βελτιώσουμε τα μέτρα εσωτερικής ασφάλειας όπως ε, καλύτερη παρακολούθηση των τρομοκρατικών ε, δραστηριοτήτων στο ίντερνετ, τα PNR για τους, ε, τα στοιχεία των επιβατών σε αεροπορικέ πτήσει κλπ. Και θα πρέπει σίγουρα να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα στο Ιράκ, στη Λιβύη και στη Συρία. Κύριε Τάνοκ, δέχεστε μια μπλε κάρτα από τον κύριο Γιάκοβτσιτς. Μάλιστα, Πρόεδρε, δέχομαι. Κύριο Γιάκοβτσιτς. Ευχαριστώ που δέχτηκεστε την μπλε κάρτα μου. Θα ήθελα να σας ρωτήσω, συμφωνείτε μαζί μου ότι μία από τις ε, χώρες που βρίσκεται σε πολύ ε, επισφαλή κατάσταση στην Ευρώπη είναι η Βοσνία Αρζεγοβίνη Εκεί έχουμε πολλούς μουσουλμάνους που αποτελούν θύματα επιθέσεων ή και υποψήφια θύματα στρατολόγηση. Δεν θα έπρεπε η Ευρωπαϊκή Ένωση να είναι ιδιαίτερα ευαίσθητη για την κατάσταση στη Βοσνία Ερζεγοβίνη. Uh, thank you Κύριο Στάνοκ, ευχαριστώ για αυτήν την ερώτηση. Ε, ενδιαφέρομαι ιδιαίτερα στα, στην περιοχή των Δυτικών Βαλκανίων. Είμαι για το Μαυροβούνιο. Παρακολουθώ πολύ στενά ε, την κατάσταση τη Βοσνία Ζεγοβίνη ω και ο συγητή, Όλε αυτέ οι χώρε των Δυτικών Βαλκανίων έχουν μουσουλμανικέ μειονότητε. Στο Κωσυφοπέδιο, για παράδειγμα, Αλβανία, Μακεδονία, Βοσνία Ζεγοβίνη. Εκεί υπάρχει σοβαρό πρόβλημα παστικοποίησης. Ε, πολλοί μαχητές της Τζιχάτ φεύγουν από εκεί. Αρκετές εκατοντάδες ε, πολεμούν αυτή τη στιγμή στις τάξεις του Ισλαμικού στρατού στο Ιράκ και τη Συρία αυτή τη στιγμή. Ε, το ΝΑΤΟ παίρνει πολύ στα σοβαρά αυτή την απειλή και θα πρέπει πραγματικά να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να αποφύγουμε αυτή τη φυγή. Thank you. Πρόεδρος, ευχαριστώ. Εκ μέρους των φιλελευθέρων, ε, κ. Μάουρα Μπαραντιαράν. Πρόεδρε, οι απόπειρες 26 Ιουνίου άφησαν πάνω από 60 νεκρούς μεταξύ αυτών και αρκετοί Ευρωπαίοι πολίτες ε, που δολοφονήθηκαν στις παραλίες της Τινησίας. Ε, αυτές οι τρεις επιθέσεις προστίθενται σε ένα ολόκληρο κύμα επιθέσεων, βίων επιθέσεων, ομών επιθέσεων, ε, μια κλιμάκωση την οποία δεν πρέπει να δεχτούμε. Ε, θα επιστρέψουν και θα χτυπήσουν ξανά, ιδιαίτερα χώρες όπως την, την που προσπαθούν να κάνουν πρόοδο στην, στο δημοκρατικό μονοπάτι και ε, οι τρομοκράτες προσπαθούν να το αποφύγουν. Εδώ πέρα Παλιότερα είχαμε πει ότι η κατάσταση της Βορειάς Αφρικής ε, πρέπει να είναι προτεραιότητα της εξωτερικής μας πολιτικής. Ε, μετά την ε, επίθεση του Εθνικού Μισό του Λμπάρδο καταλάβαμε ότι χρειάζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση με όλα τα μέσα που διαθέτει να συμμετάσχει στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας στη Βόρεια Αφρική και να βοηθήσει την Τινησία, την Αργελία, το Μαρόκο και τις άλλες χώρες της Βόρειας Αφρικής την τελευταία συζήτηση ακούσαμε πολλά για αυτό το θέμα, αλλά τι πρόοδο έχουμε κάνει, ποιοι είναι οι στόχοι που πετύχαμε, τι άλλαξε η, στην, η, η, βελτίωση οικονομίας δεν αρκεί. Εγώ θα πρέπει να επιμείνω στην ανάγκη να μπούμε ενεργά ε, στην, ε, στον αγώνα αυτό, όχι μόνο με λέξεις μια για πάντα θα πρέπει να πούμε ότι τα σύνορά μας είναι στη Βόρεια Αφρική. Δεν είναι δυνατόν να επιτρέψουμε ούτε καν ούτε ε, μια αιστεία α, αστάθειας εκεί πέρα. Δεν είναι δυνατόν να πέσει την Ισία διότι το Ισλαμικός στρατός χτυπάει την πόρτα της Ισίας και τη δική μας πόρτα. Θα ε, πρέπει να αναθεωρήσουμε την πολιτική γειτονία μα, θα πρέπει να συνεργαστούμε για την εξασφάλιση τη ασφάλεια των συνόρων μα. Δεν μπορούμε να περιμένουμε άλλο. Θα πρέπει να βοηθήσουμε ολιστικά αυτές τις χώρες που χρειάζονται τη βοήθειά μας απελπισμένα. Ε, παρ' όλα αυτά, και το επαναλαμβάνω, πάλι φοβάμαι ότι θα φτάσουμε πολύ καθυστερημένα σε αυτό το στόχο. Ευχαριστώ πολύ, Από την GUE ε, NGL το λόγο έχει η κυρία Κορνιλία Ένστ. Ένα μισή λεπτό. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Οι φρικτές επιθέσεις των τελευταίων εβδομάδων έχουν συγκλονίσει όλους μας. Αλλά νομίζω ότι έχουμε ήδη συζητήσει πάρα πολλά πράγματα για αυτή την υπόθεση και τίποτα δεν έχει αλλάξει. Ποια είναι η, η απάντηση, περισσότερη καταστολή, περισσότερη παρακολούθηση, περισσότερα κατασταλτικά μέτρα. Τι έχει φέρει όλο αυτό, τίποτα απολύτως. Πώς μπορούμε όμως να βοηθήσουμε τις χώρες αυτές όπου υπάρχει τρομοκρατία να εμποδίσουμε την στρατολόγηση τρομοκρατών. Πώς μπορούμε να ενισχύσουμε τις δημοκρατικές διαδικασίες στις χώρες αυτές. Αυτό είναι το πραγματικό ερώτημα για το Ιράκ. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτό το ερώτημα. Γιατί είναι τόσο ισχυρό το Ισλαμικό κράτος. Προφανώς έχει υποστήριξη από ένα τμήμα του πληθυσμού. Και θυμήθηκα όταν μας είπε ο επίσκοπος του Αρμπίλ ότι χρειαζόμαστε όχι όπλα αλλά υποστήριξη για την συμφιλίωση με τους Σουνίτες στον πληθυσμό. Έτσι θα μπορέσουμε να ξεπεράσουμε το πρόβλημα της τρομοκρατίας. Δεν κάνουμε τίποτα λοιπόν, δεν κάνουμε ποτέ καμία σοβαρή συζήτηση για το λόγο για τον οποίο οι νέοι πηγαίνουν και μπαίνουν σε τρομοκρατικές οργανώσεις. Θα πρέπει να καταλάβουμε και ποια είναι τα προβλήματα και οι ελλείψεις στην συμβίωσή μας και γιατί αυτοί οι νέοι τελικά απογοητεύονται και πηγαίνουν και εντάσσονται σε τρομοκρατικές οργανώσεις. Θα πρέπει να καταλάβουμε λοιπόν πού έχουμε προβλήματα σε κοινωνικό επίπεδο, τι θα μπορέσουμε να κάνουμε και δεν νομίζω ότι το PNR για τους αεροπορικούς επιβάτες θα μας προχωρήσει ούτε ένα χιλιοστό προς τη λύση αυτού του προβλήματος, απλώς θα είναι σπατάλη χρημάτων. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ακολουθεί από την ομάδα ο κύριος Νούταλ από το EFTD για τέσσερα λεπτά. Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, πριν από 15 μέρες σας είχα προειδοποιήσει ότι η επόμενη απειλή ε, δεν θα είχε ένα δυνητικό «ή» αλλά «που». Και 48 ώρες μετά είχαμε τον αποκεφαλισμό ενός ομήρου, την, τον βομβαρδισμό ενός τεμένου στο Κουβέιτ και την τρομοκρατική ε, βία στη, σε μια παραλία στη Σούς, στη Τινησία. Άρα βλέπουμε ότι όλες αυτές οι τρομοκρατικές ενέργειες είχαν κάτι κοινό, ότι γίναν εξ ονόματος του Ισλαμισμού. Υπάρχουν άλλοι στη χώρα μου που λένε ότι αυτές οι επιθέσεις δεν έχουν καμία σχέση με το Ισλάμ. Αυτό είναι γελίο αλλά και επικίνδυνο. Οι τρομοκράτες επιτελούν αυτές τις ομότητες επικαλούμενοι το Κοράνι και λέγοντας ότι αυτές οι απλές δεν έχουν καμία σχέση με το Ισλάμ. Είναι σαν να λέμε ότι ε, η Ιερά Εξέταση δεν είχε καμία σχέση με τον καθολικισμό. Θα πρέπει λοιπόν να έχουμε το θάρρος να κατονομάζουμε την πηγή. Δεν πρόκειται για την φτώχεια και την έλλειψη εκπαίδευσης. Απλώς είναι μια οπισθοδρομική ερμηνεία του Κορανίου. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να γυρίσουμε το άλλο μάγουλο, αλλά βλέπουμε ότι δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε την μισογυνία, την ομοφοβία και τους ακριοτηριασμούς. Μιλάμε για ανταλλαγή όπλων με το πετρέλαιο και αυτό γίνεται στη Σαουδική Αραβία και το Κατάρ. Θα πρέπει να πούμε πια ότι αρκεί. Διαφορετικά φοβάμαι ότι θα έχουμε να κάνουμε με μία ρήξη πολιτισμών κάποια στιγμή μέσα σε αυτό τον αιώνα και αυτό δεν θα γίνει στις ε, ρήμους της Μέσης Ανατολής αλλά στους δρόμους και τις πόλεις της Ευρώπης. Εμείς είμαστε η σημερινή πολιτική και έχουμε ένα καθήκον να δώσουμε μια καλύτερη κοινωνία στους απογόνους και δεν μπορούμε να μιλάμε για μία κοινότητα όπου πλήττονται οι ομοφιλόφιλοι και όπου υπάρχουν ε, πολίτες δεύτερης κατηγορίας. Οι χριστιανοί και οι μουσουλμάνοι είναι ίσοι. Διαφορετικά θα φανεί ότι αφήσαμε την ε, ελεύθερη και φιλελεύθερη ε, δύση σε κάτι το πιο σκοτεινό δεν μπορούμε να εθελοτυφλούμε. Πρέπει να δράσουμε. Το χρωστάμε στα παιδιά μας. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Εξ ονόματος της ε, ε, ομάδα της Ευρώπης των Εθνών για την Ελευθερία, ο κύριος Μποργέζιο. Μα εσείς θεωρείτε ότι θα αντιμετωπίσετε την Ισλαμική τρομοκρατία με αυτό το συνονθήλευμα μέσων που τα περισσότερα αργούν. Στο Συμβούλιο δεν γίνεται λόγος για σύνδεση τρομοκρατίας και παράνομης μετανάστευσης. Ο πρόεδρος της Eurojust όμως αναγνωρίζει ότι οι παράνομοι μετανάστες μπορούν να φιλτράλουν και μέλη του ίσης μέσα στην Ευρώπη. Θα πρέπει λοιπόν να μην νομιμοποιήσουμε το ακραίο Ισλάμ μέσω των ε, ε, τεμενών και των ημάμιδων. Θα πρέπει να κλείσουμε τα ακραία τεμένη, όπως θέλει να κάνει η Τινησία. Δεν μπορούμε να μιλάμε για Ισλαμοφοβή. Στο Σαρλί Επτό μίλησα με τους ανθρώπους μετά από την απαράδεκτη τρομοκρατική ενέργεια. Κανένας δεν μίλησε για Ισλαμοφοβία εκεί. Αυτός ο ε, μαζοχιστικός αντιισλαμισμός είναι η κερκόπορτα για να μπει ένα μικρόβιο το οποίο ήδη υπάρχει στην Ευρώπη. Υπάρχει μεγάλος φόβος τον οποίο ενσταλάσουμε και στην Ήπειρό μας. Γι' αυτό θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε τους τζιχαντιστές μέσα στα πλαίσια της ατζέντα μας, διότι θέλουν να επιβάλλουν τον, τον νόμο της ε, Σαρία. Ε, ξύπνησε επιτέλους ε, Ευρώπη. Ευχαριστούμε τον κύριο Μπορκέζιο. Ο κύριος Γκόλνης έχει το λόγο για ένα λεπτό. Κύριε Πρόεδρε, υπάρχουν τουλάχιστον τρία αίτια της τρομοκρατίας που εξαρτώνται από εμά. Το ένα είναι η καταστροφή, η προσπάθεια καταστροφής των κοσμικών αυταρχικών ίσως καθεστώτων τα οποία είχαν εμποδίσει την άνοδο των ριζοσπαστών. Η Λιβύη, η Συρία και η... το Ιράκ είχαν αυτή την κατάσταση. <coughs> Αυτά έγιναν με πολέμους καταστροφής από τη Δύση, με ένα αποκλεισμό ο οποίος οδήγησε σε ένα τεράστιο μίσος κατά της Δύσης. Δεύτερος αίτιο είναι η ε, παρανόηση των επιθετικών στοιχείων μιας θρησκείας όπου πολλοί θεωρούν ότι ο πόλεμος είναι ένα θεμητό μέτρο για να επεκταθεί η θρησκευτική κοινότητα και έχουν μια συγκεκριμένη στάση κατά των λεγόμενων κιαφίρ, κατά των απίστων, ακόμα και ανεάμαχοι, για να μπορέσουν να τους προσελκύσουν. Και τρίτον, είναι η μετανάστευση χωρίς κανένα έλεγχο που έρχεται από τις μουσουλμανικές χώρες και δημιουργεί μια, ένα στρώμα νέων που δεν έχουν καμία ενσωμάτωση σε μια κοινωνία και οι οποίοι είναι απόλυτα απογοητευμένοι από τον ματεριαλιστικό κόσμο και από τις σεξουαλικές ε, πρακτικές οι οποίες ξεπερνούν το φυσιολογικό. Από αυτό το έφορο έδαφος διατρέφεται η τρομοκρατία, δεν είναι όλοι αυτοί τρομοκράτες, αλλά έχουν γίνει χωρίς να το θέλουν ίσως συνένοχοι των τρομοκρατών οι μετανάστες. Ευχαριστώ πολύ, λέει Κυρία Μετσόλα, έχει το λόγο για δύο λεπτά. Ευχαριστώ. Η Ευρώπη επισκιάστηκε από την τρομοκρατία εδώ και αρκετό καιρό. Έχουν περάσει δέκα χρόνια μετά τις ιδεχθείς ε, τρομοκρατικές ενέργειες στο Λονδίνο και ε, μετά τις, τους πυροβολισμούς ε, σε μια εκκλησία στο Τσάρλεστον και το Σαρλί Εμπντό. Και η Μπόκο Χαράμ ε, προέβαλε τρομοκρατικές ε, ενέργειες, προέβησε τρομοκρατικές ενέργειες στην Ιγυρία και στην Κένια. 66 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε μία μέρα, ανεξάρτητα από τις πολιτικές τους πεπιθήσεις στη Γαλλία, το Κουβέιτ και την Τινησία. Αυτό δείχνει ότι το προσωπείο της τρομοκρατίας δεν γνωρίζει σύνορα και χρησιμοποιεί την ε, τρομοκρατία, μάλλον τη θρησκεία, ως ε, κάλυμα για τα ομά αυτά εγκλήματα. Θα πρέπει λοιπόν να μην δεχτούμε αυτή την παράλογη βία, διότι δεν εκπροσωπεί ούτε το Ισλάμ, ούτε κάποιο κράτος που είναι διεθνώς αναγνωρισμένο. Θα θέλαμε να ποτίσουμε φόρο τιμή στα θύματα της Τινησίας. Βλέπουμε ότι η Αραβική Άνοιξη ε, στην ουσία δεν μπορεί να αντιμετωπίσει την τρομοκρατία. Αυτό αφορά και την Μπόκο Χαράμ και την Αλ Σαμπάμπ. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρχει σωστή προστασία όλων των πολιτών. Είναι, ήρθε πια η ώρα να προχωρήσουμε και να αντιμετωπίσουμε την τρομοκρατία έτσι ώστε να χρησιμοποιήσουμε την ε, νομοθεσία για να αποστείλουμε ένα σαφές ε, μήνυμα από το σώμα αυτό ότι δεν θα μας φοβήσουν. Δέχεστε μία μπλε κάρτα από τον κύριο Λεμπρετών. Ωραία. Κύριε Λεμπρετόν, έχετε το λόγο. Με μικρόφωνο. Ευχαριστώ αγαπητοί συνάδελφε είπατε αναφερόμενοι στις τρομοκρατικές ενέργειες της Τινησίας, Γαλλίας και Κουβέιτ ότι θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε τη τρομοκρατία και να φτάσουμε σε μια συμφωνία. Ε, πέρα από το PNR όμως δεν μας προτείνεται τίποτα το συγκεκριμένο. Αυτό με απασχολεί κάπως, διότι δεν ξέρω κατά πόσο το PNR είναι αποτελεσματικό. Νομίζω ότι δεν είναι ένα ικανοποιητικό μέσο. Έχει έχετε συγκεκριμένες προτάσεις για την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας. Ευχαριστώ. Δεν μπορώ να, σας, να συμφωνήσω μαζί σας ότι τα μέτρα τα οποία έχουν προταθεί δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν καθόλου κατά της ε, τρομοκρατίας και των τρομοκρατών που απειλούν την ασφαλεία μας. Έχουμε πολλά μέτρα που ως ε, Κοινοβούλιο του επόμενους μήνες μπορούμε να συμφωνήσουμε. Θα πρέπει να ενισχύσουμε τον συντονιστή κατά τη τρομοκρατία, για παράδειγμα. Θα πρέπει να του δώσουμε περισσότερε ε, εξουσίες, όπω και περισσότερες εξουσίες και στην Europol, για να ενισχύσουμε τη συνεργασία ανάμεσα στι χώρε μα. Παρ' όλα αυτά, θα πρέπει να συμφωνήσουμε πρώτα μεταξύ μα. Πρόεδρος, ευχαριστώ. Ο λόγος τώρα στην κυρία Σιλβίκη Γιώμ. μισή λεπτό. Η Γαλλία, Σομαλία, Κουβέιτ, την Ισία σε μερικές ε, ώρες μόλις χτύπησε η τρομοκρατία. Είναι συντονισμένες αυτές οι ενέργειες, είναι προφανές αυτό. Έχουμε πολλές απειλές και θα πρέπει να θυμόμαστε τις παλιότερες ε, τρομοκρατικές ενέργειες αλλά χωρίς ε, ψύχωση. Θα πρέπει να ενισχύσουμε την διεθνή και την ευρωπαϊκή συνεργασία. Μόνο έτσι μπορούμε να κερδίσουμε μέσω της κοινής ευθύνης το, οι αιτίε τη τρομοκρατία είναι κοινωνικέ, οικονομικέ, ψυχολογικέ, γεωπολιτικέ κλπ. Συνεπώ χρειαζόμαστε μια ολιστική λύση. Και η σημερινή κρίση αλλάζει συνεχώ, γι' αυτό το λόγο πρέπει και εμεί να αλλάζουμε το σύστημά μα συνεχώ. Χρειάζεται να σκεφτούμε ποια είναι τα κατάλληλα μέσα για να αντιμετωπίσουμε αυτή την τρομοκρατική τζιχάντε. Ναι, χρειαζόμαστε μια αντιμετώπιση, μια επίθεση εναντίον των οικονομικών χρηματικών ροών. Θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε όλα τα μέσα που διαθέσουμε για να παρεμποδίσουμε την κυκλοφορία μέσα και έξω από το Σέγγεν των τρομοκρατών ε, τζιχαντιστών. Χρειαζόμαστε και μέτρα πρόληψης της ριζοσπαστικοποίησης η ανισότητα, η περιθωριοποίηση, ο κοινωνικό αποκλεισμό, η δυσκολία πρόσβαση στην ανώτατη εκπαίδευση, όλοι αυτοί είναι παράγοντε ριζοσπαστικοποίηση. Η Κομισιόν πολύ σωστά είπε στο πρόγραμμα, τα είπε όλα αυτά στο πρόγραμμά τη. Η παιδεία, η συμμετοχή των νέων, ε, ο διαθρησκευτικό διάλογο, όλα αυτά έχουν να παίξουν σημαντικό ρόλο στην πρόληψη τη ριζοσπαστικοποίηση. Ευχαριστώ. Ε, Ευχαριστώ. κύριος Δεμέρσμακερ έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Στις 27 ε, Ιουλίου ε, ο τρόμος χτύψε τη Γαλλία, την, την, την Ισία, το Κουβέιτ, αλλά και την Νιγηρία. ε, ε αθώοι, τουρίστες, πιστοί, απλοί πολίτες χτυπήθηκαν και έχασαν τη ζωή τους. Δεν θα πρέπει να επιτρέψουμε στον εαυτό μας ε, να μας, αποσπάσει, ε, να μας αποσπάσουν αυτές οι ενέργειες από το στόχο μας. Ε, στην Τινησία ξεκίνησε η Αραβική Άνοιξη. Η κοινωνία εκεί όμως είναι πολύ ευάλωτη και οι τρομοκρατικές αυτές επιθέσεις πλήττουν και τον τουρισμό. Η Τινησία χρειάζεται μέλλον. Αυτή η ιδέα του μέλλοντος είναι πολύ σημαντική. Θα πρέπει να τη δουλέψουμε. Ας σκεφτούμε ένα, Marshall Plan, ένα σχέδιο Marshall ε, μέσω μιας περιφερειακής ε, συνεργασίας. Ε, θα πρέπει να βοηθήσουμε και τη Νέα Λιβύη ε, για να μην τη χάσουμε υπέρ του ISIS, του Ισλαμικού στρατού. Ευχαριστώ κυρία Γκρίσμπεκ. Ένα λεπτό. Ε, απέναντι στην τρομοκρατική απειλή θα πρέπει να μας ενώνουν όχι μόνο τα ε, λόγια αλλά και οι δράσεις και τα μέσα για να προστατέψουμε τις αξίες μας, τους πολίτες μας και να προλάβουμε αυτές οι δεχθείς ε, πράξεις τις οποίες, των οποίων είμαστε μάρτυρες θα πρέπει να δείξουμε αυστηρότητα για στην τρομοκρατία διότι εκεί διακυβεύεται η δημοκρατία μας. Πρόληψη της ροσπαστικοποίησης, παρακολούθηση των δικτύων που χρησιμοποιούνται από τους τρομοκράτε για την προπαγάνδα τους, την οσυρή του προπαγάνδα, ιδιαίτερα ε, για τους νέου Η καταπολέμηση του λαθρεμπορίου των όπλων πρέπει να είναι προτεραιότητα και χαίρομαι που ο Λουξεμβούριο Υπουργό τα ανέφερε. Θα πρέπει όμω να ενώσουμε τι προσπάθειές μα στην ανταλλαγή πληροφοριών και στο συντονισμό της. Θα πρέπει να πολλαπλασιαστεί η ανταλλαγή πληροφοριών και θα πρέπει να γίνει υποχρεωτική βέλτιστοποιώντας την Europol και δημιουργώντας ένα πραγματικό ευρωπαϊκό PNR που θα πρέπει να είναι αποτελεσματικό. Θα πρέπει να ε, μεταρρυθμιστεί το SIS ε, για, σε ό,τι αφορά ιδιαίτερα τις προειδοποιήσεις ε, για τους ύποπτους τρομοκρατίας. Η κοινή πολιτική ασφάλειας είναι απόλυτος απαραίτητη και το ζητούν οι πολίτες μας. Μάιερ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κοιτάξτε, είναι πραγματικά τρομακτικό και δεν χρειάζεται να ανατρέξουμε βαθιά στο παρελθόν για να δούμε ουσιώδεις αλλαγές στην κοινωνία μας. Η Τινησία, η Γαλλία και πάλι η Γαλλία, το Κουβέιτ. Εγώ έρχομαι από το Γκράτς της Αυστρίας όπου πριν από τρεις εβδομάδες έλαβε χώρα μία επίθεση με τρεις νεκρούς και 40 τραυματίες και δεν ήταν σαφές κατά πόσον και αυτό δεν είχε πραγματοποιηθεί από έναν Ισλαμιστή. Βεβαίω, αυτά όλα είναι ιδιαίτερα τρομακτικά και ιδιαίτερα τρομακτικά ή τρομακτικό είναι το γεγονό ε, πώ ε, ε, αντιμετωπίζει κανεί αυτή την κατάσταση. Πολλοί προειδοποιούν ότι αυτό το ριζοσπαστικό Ισλάμ δεν θα φοβηθεί και να δραστηριοποιηθεί στην Ευρώπη. Προειδοποιούμε ότι το ριζοσπαστικό Ισλάμ είναι μέσα στην κοινωνία μα και διαβάζουμε συνεχώ σε μέσα ενημέρωση και σε υπεύθυνου πολιτικού ότι αυτά είναι μεμονωμένε περιπτώσει και σιγά σιγά εγώ έχω την εντύπωση ότι εδώ έχουμε να κάνουμε με στρατό των ε, ε, φυτών. Και υπάρχουν τρεις ε, δρόμοι που είναι πολύ επικίνδυνοι. Εκεί λοιπόν δραστηριοποιούνται οι καμικάζοι. Το επόμενο πεδίο μάχης θα είναι η Ευρώπη, αυτό λέει ο κόσμος, και λόγω της, της ε, ροής των μεταναστών και λόγω της αποτυχίας ε, των κυβερνήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης αυτό είναι ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα με τα οποία θα πρέπει να ασχοληθούμε τα επόμενα χρόνια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο Τζοντ Πάτον. Δύο λεπτά. Α, όχι, εσείς όμως πήρατε το λόγο πριν. Καλά, ξαναπάρτε τον άντε. Ο συνάδελφός μου Πολ Νάτσελ που μίλησε πριν από λίγο είπε πολλά από αυτά που ήθελα να πω και εγώ και με τα οποία φυσικά συμφωνώ. Η απειλή που αντιμετωπίζουμε όλοι εδώ στη Δύση και όχι μόνο προέρχεται από το ριζοσπαστικό Ισλάμ. Οι εξτρεμιστές έχουν ένα κοινό χαρακτηριστικό. Διαβάζουν όλοι το ίδιο βιβλίο, το Κοράνι το οποίο περιλαμβάνει εκκλήσεις όπως σκοτώστε τους απίστους όπου τους βρείτε. Τρομοκρατήστε τους άπιστους και μερικοί αυτά τα παίρνουν κατά γράμμα. Μας λένε, τους λένε οι ηγέτες τους ότι το Ισλάμ είναι θρησκεία ειρήνης και αγάπης, αλλά αυτό δεν συμβαδίζει πολύ με το κείμενο. Το πρόβλημα είναι ότι η εξτρεμιστές ε, έχουν δίψα για αίμα και νομίζουν ότι έτσι θα πάνε πιο γρήγορα στον παράδεισο. Οι δυτικές φιλελεύθερες δημοκρατίες πρέπει να καταλάβουν ότι το εξτρεμιστικό και ζηλωτικό Ισλάμ δεν έχει καμία θέση στην κοινωνία μας. Έχω γνωρίσει και εγώ κάθε μέρα συναντάω φιλιρινικούς μουσουλμάνους τους οποίους πρέπει να υποστηρίξουμε έναντι των εξτρεμιστών. Ο Σούντσου είπε ο πόλεμος κερδίζεται πρώτα στο μυαλό του αντιπάλου και πρέπει να καταλάβουμε τη δύναμη του λόγου. Αν ελέγξουμε το λόγο της λέξης θα μπορέσουμε να νικήσουμε. Ο χριστιανισμός, ο βουδισμός, ο Ιουδαϊσμός είναι γνωστές ως φιλιρινικές θρησκείες αλλά το Ισλάμ το δεχόμαστε ως ακραίο. Παλιά το λέγαμε Μωαμεθανισμό γιατί είναι η θρησκεία του Μωάμεθ όπως ο Βουδισμός είναι η θρησκεία του Βούδα κτλ. Λοιπόν πρέπει να εξηγήσουμε ότι αυτή την ιδεολογία δεν τη δεχόμαστε και πρέπει να πάρουμε πρακτικά μέτρα για να κερδίσουμε τον πόλεμο κατά των ακραίων αυτών ανθρώπων αν θέλουν να ζήσουν υπό τον νόμο της Σαρίας πάνε σε κάποια άλλη χώρα όπου μπορούν να τον εφαρμόσουν. Η κυρία Τερέζα Χιμένες Μπεσερίλ Μπαριό. μισή λεπτό, παρακαλώ. Ε, Πρόεδρε, τα πρώτα λόγια μου θέλω να είναι για τα θύματα στα οποία αφιερώνω τη δουλειά μου όλοι εδώ. Πάντα υποστήριξα ότι στο Κοινοβούλιο πολλοί είμαστε αυτοί που θυμόμαστε την τρομοκρατία μόνο όταν υπάρχει επίθεση. Και όταν, ε, όταν περάσει, περάσουν οι ειδήσει ξεχνιούνται. Δυστυχώ αυτή η απειλή υποτιμήθηκε ε, για πολύ καιρό και τώρα έγινε κάτι πολύ σοβαρό που τρομοκρατεί την κοινωνία μας. Αυτό είναι η νίκη των τρομοκρατών. Σκοτώνουν ένα για να φοβήσουν όλους και να πάψει έτσι να υπάρχει ελευθερία μας. Δεν χρειάζεται να ταξιδέψουμε στο, στην Τίνιδα, στο Παρίσι, στο Λονδίνο. Αυτοί μπορεί θέλησαν να, ε, να σπείρουν το φόβο στο κέντρο της Ευρώπης. Γι' αυτό χαίρο που η Προεδρία του Λουξεμβούργου θεώρησε ως προτεραιότητά της τη μάχη κατά της δημοκρατίας. Ζητώ να μπει το θέμα στο θέμα ασφάλειας καλύτεροι μηχανισμοί προστασία γιατί είναι ο καλύτερος τρόπος να αντιμετωπίσουμε αυτού που θέλουν να καταστρέψουν το πλέον ιερό των δικαιωμάτων, το δικαίωμα στη ζωή. Θέλω να στείλουμε ένα σαφές μήνυμα στους τρομοκράτες. η κοινωνία μας με χρόνια κοινέ αξίες δεν θα ε, υποχωρήσει στα μαχαίρια, στις βόμβες και στα όπλα. Υποστηρίζω τη μνήμη των θυμάτων γιατί με αυτόν τον τρόπο προστατεύω και υπερασπίζομαι την αξιοπρέπεια όλων των Ευρωπαίων που ουδέποτε, ουδέποτε θα παραχωρήσουμε την ελευθερία μας. Θυμίζω σε πολλούς εδώ στο σώμα ότι η ελευθερία δεν, είναι, δεν χωρίζεται από την έννοια της ασφάλειας. Ευχαριστώ. Δέχεστε μια μπλε κάρτα από την κυρία Νταϊάννα Ντότζ. Δέχεστε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ την κυρία Βουλευτή για αυτά που είπε και ιδιαίτερα για όσα έχει κάνει για τα θύματα της τρομοκρατίας συμφωνεί ότι πρέπει να στηρίξουμε τα θύματα αυτά και να διασφαλίσουμε ότι το Κοινοβούλιο και οι κυβερνήσεις μας θα κάνουν σαφή διαχωρισμό και νομοθετικά μεταξύ εκείνων που διαπράττουν τρομοκρατικές ενέργειες από τη μία και τα αθώα θύματα από την άλλη. Βεβαίως. Ευχαριστώ πολύ για την ερώτησή σας. Νομίζω ότι ήρθε η ώρα να γίνει ένα ψήφισμα για τα δικαιώματα των θυμάτων της δημοκρατίας ποτέ δεν είναι ίδιος ένας άνθρωπος που που δέχεται μια σφαίρα στην πλάτη της. Εδώ έχουμε να συζητήσουμε όχι μόνο την Ισλαμική τρομοκρατία, πρέπει να συζητήσουμε την τρομοκρατία της ΕΤΑ που σκοτώνει επίσης τα θύματα της. Το πρόβλημα είναι ότι λείπει μια σαφή ιδέα. Εσείς και εγώ μπορεί να το έχουμε σαφές στο μυαλό μας. Πολλοί δεν έχουν ωστόσο στο μυαλό τους τι χρειάζεται. Χρειάζεται νομοθεσία διότι τα θύματα της τρομοκρατία είναι εκπρόσωποι κάθε τμήματο τη κοινωνία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ο κύριος Βάντερ Χόλτς, ένα, ένα λεπτό. Δυστυχώς ε, βλέπουμε ότι έχουμε όλο και περισσότερα αθώα θύματα ε, των επιθέσεων και αυτό το βρίσκω πολύ απειλητικό. Φοβάμαι ότι αυτή δεν θα είναι η τελευταία φορά αλλά ότι τέτοιου είδους καταστάσεις θα έρχονται και θα επανέρχονται. Απλά μπορούμε να ελπίζουμε ότι ε, θα έχουμε μεγαλύτερα διαλύματα. Ο εχθρός είναι ένας ε, πολύ αρνητικός εχθρός και έχει πολιτισμό μας, ε, την ελευθερία, την ελευθερία απόψή την ανεξιθρησκεία, το πώς θέλουμε να ζούμε. Αυτό λοιπόν τον εχθρό πρέπει να τον αντιμετωπίσουμε με όλα τα απαραίτητα μέσα, με ξυπνάδα, αποφασιστικότητα και προδραστικότητα. Πρέπει λοιπόν να ε, αντιμετωπίσουμε το ριζοσπαστικό τρόπο, πρέπει να μπούμε μέσα στα δικά τους, στους δικούς τους τους κύκλους και πρέπει να αναζητήσουμε τα αιτία γιατί οι άνθρωποι πέφτουν στα δίχτυα αυτών των τρομοκρατών και αυτόν τον αγώνα πρέπει να τον κερδίσουμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κίκ Χοπ, ένα λεπτό παρακαλώ. Τιμωθή Κίκ Χοπ. Πρόεδρε, συμφωνώ με αυτά που υπόθηκαν για την τρομερή επίθεση στην Τινησία που δείχνει πόσο ευάλωτοι είναι όλοι οι άνθρωποι εναντίον ενός αποφασισμένου εχθρού. ε, όλες αυτές οι τελευταίες επιθέσεις δείχνουν ότι είμαστε ευάλωτοι παντού. Δεν είναι τρο, φόβ, φόβος απλώς, είναι πραγματικότητα. Και η πραγματικότητα αυτή ξεπερνάει τα δικά μας σύνορα. Είναι ζωτικό λοιπόν να συνεργαστούμε και με τρίτες χώρες για να διασφαλίσουμε την ασφάλειά μας και φυσικά μια αποτελεσματική στρατηγική και για την ανταλλαγή πληροφοριών. Η Τινησία όπως και άλλες χώρες και στην Ευρώπη δεν μπορούμε να περιμένουμε ότι η Τινησία θα ανταποκριθεί μόνη της, θα αντιμετωπίσει μόνη της αυτή την απειλή. Χρειαζόμαστε μια ενιαία στρατηγική για να καταπολεμηθεί το λεγόμενο Ισλαμικό κράτος και η τρομοκρατία. Ευχαριστούμε. Αυτή τώρα. του Αρουής, η κυρία Ατουντού Αρουής. Ευχαριστώ πρόεδρε. Η μάχη κατά του Ισλαμικού, του, το, της Ισλαμικής δημοκρατίας θα χαράξει τον 21ο αιώνα. Πρέπει να είμαστε ωστόσο αποφασικοί. Πρέπει να χτυπήσουμε την νομιμοποίηση με, με αποτελεσματικότητα ο λόγος είναι εξίσου σημαντικός με τη μάχη. Πρέπει να μας ε, ακολουθήσει και η κοινωνία. Δεν υπάρχουν ασφαλή σύνορα. Πρέπει να εμπλακούμε σε όλο το πλανήτη, προστατεύοντας κάθε πολίτη που θέλει να είναι ελεύθερος. Άρα πρέπει να έχουμε σαφή εικόνα. Κύριε Επίτροπο, για να, για να είμαστε ηγέτες της κοινωνίας πρέπει να είμαστε γενναίοι. Ταυτόχρονα χρειαζόμαστε να παγιώσουμε, να ενισχύσουμε τη δημοκρατία εκτός Ευρώπης. Η τωρινή γεωστρατηγική κατάσταση, η συμμαχία με ηγέτες που δεν είναι πάντα δημοκρατικοί, σίγουρα θα πάψουν να είναι αποτελεσματικές μορφές συνεργασίας βραχυπρόθεσμα. Πάντως, τη μάχη αυτή έχετε την υποστήριξή μας γιατί είναι κάτι ζωτικό για όλους μας. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ο δικός μας ο εχθρός ε, δεν είναι ένας, δεν μπορούμε να τον εντοπίσουμε. Έχουμε τους εχθρούς ολόκληρο τον κόσμο. Δεν έχει πρόσωπο, δεν βρίσκεται σε ένα συγκεκριμένο σημείο, αλλά ε, έχει μπει στην καθημερινότητά μας, ε, επιτίθεται σε εργοστάσια, σε παραλίες. Ο δικός μας ο εχθρός δεν υπερασπίζεται μία συγκεκριμένη χώρα, ούτε μία οικογένεια, αλλά μία έννοια, μία άποψη την άποψη εκείνη με την οποία η θρησκεία επηρεάζει όλες τις εκφάνσεις της ζωής και η πιστή πρέπει να είναι ενωμένη. Πρέπει λοιπόν να δούμε πώς οι επιθέσεις στη Γαλλία, στη Σομαλία, στο, Κουβά, στο Κουβέιτ συντονίστηκαν. Αυτό βέβαια δεν έχει τόσο μεγάλη σημασία. Τώρα οι προκλήσεις διαδίδονται όλο και περισσότερο και γι' αυτό λοιπόν πρέπει να συνενώσουμε τις δυνάμεις μας για να καταλήξουμε σε επίγουσες και ουσιαστικές δράσεις. Δεν είναι εύκολο αυτό γνωρίζω πάρα πολύ καλά, αλλά έχω την εντύπωση ότι όταν μιλάμε για το ε, πώς θα αντιμετωπίσουμε τους τρομοκράτες τζιχαντιστές. Μπαίνουμε δυστυχώς σε πολιτικές συζητήσεις, μπλεκόμαστε σε αυτές που είναι ε, πολύ εκφοβιστικές. Ο αγώνας για την αντιμετώπιση του ρίζοσπαστισμού, της προπαγάνδας, ε, τις διάφορες στρατηγικές ε, χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, αυτά πρέπει να τα συζητάμε πιο συχνά και όλοι από κοινού να βρούμε συγκεκριμένες προτάσεις. Ο Πέρες ε, Σκιβέλ είπε ότι η μόνη ελπίδα για να αντιμετωπιστεί η τρομοκρατία βρίσκεται στην τήρηση και το σεβασμό των δημοκρατικών κανόνων. Περισσότερη δημοκρατία αλλά και ελευθερία για αυτές τις χώρες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και τώρα ο κύριος Βιώτη, η κυρία Βιώτη. Ο κύριος Βιώτη, με συγχωρείτε, Ντανιέλε Βιώτη. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δημιουργήθηκε ως δύναμη ειρήνης, ως δύναμη που θα εμποδίσει τον, τον δρόμο, το μίσο στην καταστροφή εντός και εκτός των συνόρων της. Οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν θέτουν σε κίνδυνο την συνοχή μας και αυτό είναι, επιλογή, είναι αποτέλεσμα των επιλογών των κρατών, των κρατών που κάνουν επιλογές συμμάχων χωρών εκτός της Ένωσης και της εξωτερικής τους πολιτικής. Εμείς πρέπει να έχουμε υποχρέωση να ξεκινήσουμε εκ νέου την κοινή μας δράση, κοινή δράση εξωτερική για όλη την Ένωση, με ενιαίες προσεγγίσεις για την ασφάλεια, για την αντεργή πληροφοριών, για τη συνεργασία. Πρέπει να ειδοποιήσουμε πολιτικές κοινωνικής ένταξης και να χτυπήσουμε το μίσος κυρίως το μίσος που είναι αιτία των, δραματικών γεγονότων που είδαμε τα τελευταία χρόνια στην Τινησία, στη Γαλλία και αλλού. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να βγει από την λογική της επιτήρησης και τιμωρίας. Έχουμε την ευθύνη, την υποχρέωση να σεβαστούμε κατά βάση τις θεμελιώδεις ελευθερίες των ανδρών και γυναικών σε άλλα κράτη εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και να έχουμε σαφή εικόνα του ότι η ασφάλεια δεν είναι ε, λόγος ε, καταπολέμησης της δημοκρατίας. Γι' αυτό ζητάμε από το Κοινοβούλιο να υποστηρίξει το, το όσο πιο ενεργά γίνεται την επίτροπο, την ύπατη εκπρόσωπο και αντιπρόεδρο κυρία Μογκερίνη σε αυτή την ε, στροφή προς, την κοσμική, προς τα κοσμικά κόμματα που είναι ίσως ο καλύτερος τρόπος να χτυπήσουμε την δημοκρατία. Ευχαριστώ κύριε Βιώτη. Ο κύριος Πιετρόφσκι, 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Αυτές οι τρομοκρατικές επιθέσεις ήταν πολύ βίαιες, πολύ καλά οργανωμένες ε, αρχηγοί του Ισλαμικού κράτους, ο αρχηγός ο ένας που ε, ομολόγησε αυτό το έγκλημα, είπε ότι θα γίνονται δολοφονίες ε, χωρίς ε, κανέναν διασμό, χριστιανούς, ε, τουρίστες, αυτό που ζήσαμε στην Τινησία αλλά και στη Γαλλία και αλλού, εκεί αποκεφαλίζουν τους ανθρώπους, κόβουν το κεφάλι οι πολεμιστές ε, δείχνουν την αποφασιστικότητά τους και τη δύναμή τους και η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι αμήχανη. Ε, δυστυχώς αυτό είναι ένα αποτέλεσμα της δικής μας της πολιτικής γιατί δεν ενισχύσαμε τις ΗΠΑ στον αγώνα κατά της τρομοκρατίας. Και μόνο αυτό, αλλά αποδυναμώσαμε αυτόν τον αγώνα με αυτές τις περίεργες εδώ εξεταστικές επιτραπές ε, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Υπάρχει λοιπόν μια περίεργη περιδίνηση και αυτή είναι εμείς φέραμε στο προσκήνιο. Οι τρομοκράτες ε, προστατεύονται από περίεργα ανθρώπινα δικαιώματα. Αυτή λοιπόν είναι μια λάθος πολιτική και πρέπει να την αλλάξουμε. Αυτό είναι το πρώτο βήμα για να αντιμετωπίσουμε την τρομοκρατία προς όφελος των λαών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βίκτορ Μποστινάρου. κύριος Μποστινάρου έχει το λόγο για δύο λεπτά. Τσίνκο Μπάρτζο, πρόεδρε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα, ε, πρέπει να σας πω, με εντυπωσίασαν ε, τα λόγια που είπατε και πριν ε, στα ρουμάνικα. Κύριε Πρόεδρε, πρόκειται για μια οργανωτική δομή ε, της οποίας η στόχη είναι ο προσωλητισμός και η προπαγάνδα. Αυτό είναι ο βασικός στόχος ε, των τρομοκρατών που είναι να υπονομεύουν τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δομή της κοινωνίας. Η τρομοκρατική δραστηριότητα είναι μια κοινή απειλή που αφορά όλους ε, με μια αυξανόμενη δυναμική. Είναι μόνο η αρχή του 2015 και σε παγκόσμιο επίπεδο έχουμε καταγράψει 138 τρομοκρατικές επιθέσεις από τις και 6 εξ αυτών ε, είναι από γνωστές τρομοκρατικές οργανώσεις όπως από την Ίση, την Μπόκο Χαράμ, την Αλ Σαμπάμπ ή τους ε, Ταλιμπάν. Υπάρχουν όμως και οι long δηλαδή ε, τρομοκράτες ε, που λειτουργούν μόνοι τους. επιθέσεις στην Τινησία, στο Μάλι, στην Κένια, στη Συρία, ε, στο Κουβέιτ και σε άλλες χώρες έπληξαν όχι μόνο συγκεντρωμένους ανθρώπους και τρομοκράτες αλλά και πολλούς άλλους ανθρώπους. Επίσης έπληξαν και τις δύναμης την αστυνομία για να αποσταθεροποιήσουν της ε, τα κράτη και για να υποσκάψουν την εμπιστοσύνη της ε, διεθνούς ε, κοινωνίας έναντι της δυνατότητας των κρατών να ελέγχουν αυτό το φαινόμενο. Όμως η τρομοκρατική απειλή δεν συγκρατείται, δεν σταματάει στα σύνορα. Είδαμε λοιπόν τις επιθέσεις αυτές ε, και σε άλλες χώρες. Στην Αυστρία, παραδείγματο χάρη. Και θα υπάρξουν και άλλες επιθέσεις στα κράτη-μέλη. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό να ενισχύσουμε τη συνεργασία ανάμεσα στα κράτη-μέλη για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε αυτές τις απειλές και για να έχουμε μια ολοκληρωμένη προσέγγιση ε, του στρατηγικού ε, στόχου μας. Να υπάρχει μια στρατηγική ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης Αυτά τα αποφασίσαμε στο Συμβούλιο και του Φεβρουαρίου και επαναλήφθηκαν πρόσφατα και στο Συμβούλιο του Ιουνίου. Άρα δηλαδή πρέπει για το 2016 να προετοιμάσουμε μια ε, στρατηγική για την ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ασαρκάν, επόμενος ομιλητής, ε, παρακαλώ έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε αντιμετωπίζουμε απειλές κάθε μέρα. Οι πρόσφατες τρομοκρατικές επιθέσεις του Ισλαμικού κράτους μας το δείχνουν. Δεν έχουν κανένα έλεος ούτε διαχωρίζουν μεταξύ των ανθρώπων. Είναι απλή λίσταρχη. Τις τελευταίες εβδομάδες σκότωσαν τουρίστες στην Τινησία, Αιγυπτίους στρατιώτες στο Σινά και Πακιστανούς ταξιδιώτες στο Καράτσι καθώς και αποκεφάλισαν κάποιον στη Γαλλία. Οι αριθμοί των θανάτων θυμίζουν, μας θυμίζουν ότι η καταπολέμηση του εξτρεμισμού είναι κάτι που δεν έχει τελειώσει. Υπάρχουν όμως και καλά νέα. Ο μουσουλμανικός κόσμος όλο και πιο πολύ παίρνει θέσεις στεναρά κατά των ακραίων θέσεων και των επιθέσεων στο όνομα του Ισλάμ. Η Ένωση πρέπει να υποστηρίξει τέτοιες προσπάθειες από ε, ε, κυβερνήσεις τρίτων χωρών. Παρόλα αυτά, η μακροπρόθεσμη λύση θα εξαρτηθεί από τη ε, λύση των, της ρίζας του κακού, όπως την ειρήνευση στη Μέση Ανατολή. Πρέπει για να κερδίσουμε, να κερδίσουμε τον πόλεμο κατά του εξτρεμισμού εδώ στην Ευρώπη. Σε πρόσφατη δημοσκόπηση φάνηκε ότι 46% των Βρετανών θεωρούν ότι οι μουσουλμάνοι δεν συμμερίζονται τις βρετανικές αξίες. Αυτό είναι τρομερό, γιατί όχι μόνο είναι ψέμα, αλλά δεν δικαιολογεί και τις εξτρεμιστικές τάσεις. Πρέπει λοιπόν να συνεργαστούμε με ηγέτες κοινοτήτων αν να διασφαλίσουμε ότι η κοινωνική δικαιοσύνη και η οικονομική ευημερία θα συμβαδίσουν. Ευχαριστώ. Δέχεστε γαλάζια κάρτα από τον κύριο Κάρσκι. Δέχετε. Ορίστε κύριε Κάρσκι μου. Ευχαριστώ πρόεδρε. Το ερώτημά μου αφορά την αυξανόμενη μετανάστευση από το νότο της Μεσογείου προς την Ευρώπη, τον νότο, την άλλη πλευρά της Μεσογείου. Δεν θεωρείτε ότι πρέπει να περιοριστεί αυτή η ροή ώστε οι τρομοκρατικές απειλές που μπορεί να αντιπροσωπεύει να μην φτάσουν ως την Ευρώπη. Νομίζω η καλύτερη απάντηση δεν είναι αυτή. Αυτό που χρειάζεται να γίνει είναι να δούμε τους λόγους γιατί τόσο πολλοί άνθρωποι που έχουν οικογένεια, σπίτι αναγκάζονται να φύγουν. Πρέπει λοιπόν να υπάρξει περισσότερη σταθερότητα στον κόσμο, περισσότερη ισότητα. Μόνο άμα λυθούν αυτά θα μπορέσουμε τελικά να λύσουμε και το πρόβλημα που μας απασχολεί. Όχι επιτιθέμενοι στους μετανάστας. Ευχαριστούμε. Δέχεστε κι άλλη μπλε κάρτα από την κυρία Βίνμπεργκ. Ναι. Ορίστε κυρία Βίνμπεργκ μου. Ευχαριστώ. Ακούσαμε να λένε όλοι ότι κάτι πρέπει να γίνει από τον καθένα μας. Σωστά, αλλά ποιες είναι οι προτάσεις, συγκεκριμένες προτάσεις για να σταματήσει, σταματήσει να γίνεται αυτό που γίνεται στη χώρα μου, για παράδειγμα, όπου υπάρχουν ξένοι μαχητές, στους οποίους δίνουμε δουλειά, που προσπαθούν να επανενταχθούν. Γιατί δεν υφίστανται κυρώσεις οι άνθρωποι αυτοί γιατί δεν ε, αφαιρείται η ηθαγένειά τους για να μην μπορούν να γυρίσουν ποτέ στην Ευρώπη. Απαντήστε σας παρακαλώ. Η απάντηση είναι ξεκάθαρη. Αυτοί που έχουν διαπράξει αδικήματα πρέπει να ε, φυλακιστούν. Οι αθώοι δεν θα έπρεπε να τιμωρηθούν. Κατά συνέπεια αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να έχουμε ασφαλείς πολιτικές, σίγουρες πολιτικές που θα εξασφαλίσουν ότι όσοι διέπραξαν αδικήματα κύματα δεν θα υφίστανται ατιμορρησία, αλλά ταυτόχρονα ότι αυτοί που δουλεύουν σκληρά την χάνουν ίσης αντιμετώπισης και μπορούν να συνεχίσουν να δουλεύουν σκληρά. Ευχαριστώ. Και εγώ ευχαριστώ. Ο κύριος Φουντούλης. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η Ευρώπη δυστυχώς βιώνει τον τελευταίο καιρό ένα κύμα τρομοκρατικών επιθέσεων δεκάδες άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους. οι συμπολεμιστές και συνοδοιπόροι των τρομοκρατών του ισλαμικού χαλιφάτου εισάγουν και στις πατρίδες μας τον τρόμο. δυστυχώς με το φανατισμό που τους διακρίνει και την αδυναμία των ευρωπαίων να δώσουν μια αποφασιστική απάντηση οι επιθέσεις αυτές θα αυξηθούν δραματικά στο μέλλον. η χρυσή αυγή έχει ξεκάθαρη θέση ενάντια στην τρομοκρατία. πρέπει να βρούμε τον τρόπο να θωρακιστούμε από του εισβολείς. πρέπει να δώσουμε μια ισχυρή απάντηση σε αυτέ τι άνανδρες πράξεις μπορώ και δικαιούμαι να μιλάω με οργή αλλά και πόνο. ενάμιση χρόνο πριν όταν άναδρα και ανέντιμα αριστεροί τρομοκράτες δολοφόνησαν το γιο μου γιώργο φουντούλη και το φίλο του μανώλη καπελώνη δύο νέα παιδιά μπροστά από τα γραφεία μας δεν υπήρξε καμία αντίδραση από όλους όσους παρουσιάζονται τόσο ευαίσθητοι σήμερα. ζητάω και σήμερα πάλι τη στήριξή σας ώστε η 1η Νοεμβρίου να κηρυχτεί πανευρωπαϊκή ημέρα κατά της τρομοκρατίας. Θα ήθελα να επιδεικνύει το Κοινοβούλιο την ίδια ευαισθησία για όλες τις τρομοκρατικές επιθέσεις από όπου και αν προέρχονται. κανείς από το πολιτικό σύστημα τότε δεν καταδίκασε τις επιθέσεις κανένας δεν ενδιαφέρθηκε να βρεθούν οι δολοφόνοι κάποιοι δεν ασχολήθηκαν γιατί έτσι τους συνέφερε πολιτικά. αυτό είναι κάτι που με κάνει και αναρωτιέμαι είμαστε καλύτεροι από τους τρομοκράτες ή απλά κρυβόμαστε πίσω από ένα ψεύτικο προσωπείο. σας ευχαριστώ. ευχαριστώ. Anapoliotis. Now it's time for... Η, η διαδικασία του Catch the Eye τώρα. Ευχαριστώ. Είναι ευθύνη όλων μας να προστατεύσουμε την ζωή μας, τη ζωή όλων στον κόσμο. Η τρομοκρατία δείχνει ότι μπορούμε να είμαστε θύματα παντού και πάντα. Δεν υπάρχει εξήγηση για κάτι τέτοιο. Τα γεγονότα αυτά πρέπει να αποφεύγονται. Πρέπει να συνεργαστούμε αναζητώντας εταίρους ανά τον κόσμο, όπως είπε και ο κύριος Επίτροπος. Πρέπει να διορθώσουμε τα εργαλεία που έχουμε στη διάθεσή μας και χρειαζόμαστε μορφωμένους και αποτελεσματικούς υπεύθυνους στις διοπτικές αρχές. Θέλω να μιλήσω για τα αθώα βήματα που διώκονται για τις πεπιθήσεις τους και σκέφτομαι τους χριστιανούς, συχνά παιδιά ή γυναίκες που υφίστανται τις ε, βιοπραγίες του Άισις, πέραν της απώλειας ανθρώπινων ζώων, θα πρέπει να μιλήσουμε και για τα, ε, ε, τα μνημεία που πολλές φορές είχαν ηλικία χιλιάδων ετών και που καταστρέφονται. Όλη η ανθρωπότητα χάνει από αυτό. Ευχαριστώ. Η κυρία Σουζούλικα. Ο κύριος Τζούλικα, συγγνώμη. Λόγω των τρομοκρατικών επιθέσεων, ο κόσμος στην Ευρώπη αντιμετωπίζει ένα πολύ σοβαρό κίνδυνο. Πιστεύω ότι η παγκόσμια απειλή θα πρέπει να αντιμετωπίσει την παγκόσμιο τρόπο. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο να, κάνουμε κάθε, να λαμβάνουμε κάθε μέτρο για τη διαφύλαξη της ασφάλειας των πολιτών μας και να παίξουμε έναν ρόλο στήριξη στις ε, απειλές αυτές. Οι τρομοκρατικέ απειλέ υπονομεύουν την κοινωνία και τον τρόπο ζωή μα Είναι μια απευθεία επίθεση στις βασικές αξίε της Ένωσης, του κράτους δικαίου, του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θερμοκρατικών δικαιωμάτων των πολιτών. Η ενότητα στη διαφορετικότητα και της ενότητα στη διαφορετικότητα αποτελεί απειλή στην ευημερία που προσπαθεί να παράσχει στους πολίτες της Ευρωπαϊκή Ένωση. Πιστεύω ότι η πρόληψη και η καταπολέμηση της τρομοκρατίας σημαίνει ότι η ασφάλεια και η ανθρώπινα δικαιώματα είναι συμπληρωματικά και ότι η ευρωπαϊκή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλεια αντιμετωπίσει την τρομοκρατική απειλή και τα αίτια της ανά τον κόσμο. Ευχαριστώ. Hvala lijepa. Teroristički napadi Στην ε, Γαλλία οι επιθέσεις ε, οι οποίες ε, έλαβαν χώρα δείχνουν ότι στην Ευρώπη υπάρχουν και εσωτερικέ απειλές. Οι ε, τουρίστες είναι βάλωτοι. Θα πρέπει λοιπόν να γνωρίζουμε ότι η αντιμετώπιση των Ισλαμιστών είναι πολύ ήπια, αλλά ήπιοι είμαστε και έναντι εκείνων οι οποίοι έχουν ανατραφεί μέσα στο μίσος. Σήμερα λοιπόν η Ευρώπη ε, φοβάται και ντρέπεται να προβάλλει τις χριστιανικές της αξίες, σαν να ντρέπεται να προβάλλει την ταυτότητά της. Αυτό όμως είναι πρόβλημα γιατί εμφανίζονται νέα κράτη με νέες ε, ταυτότητες. Ε, γι' αυτό λοιπόν το λόγο ε, μην ξεχνάμε ότι με τον τρόπο μας στηρίζουμε ή ευνοούμε την ανάπτυξη τέτοιων επιθέσεων. Οι επιθέσεις αυτές όμως βλάπτουν άλλους ανθρώπους και πρέπει να τους επισημάνουμε ότι δεν έχουν το δικαίωμα να διαπράττουν τέτοιου είδους πράξεις. Σας ευχαριστώ πολύ. Επίτροπε, συνάδελφοι, στα νότια σύνορα κάτω από την Ευρώπη ο αραβικός κόσμος αντιμετωπίζει σκληρές συγκρούσεις, εξαφανίζονται ολόκληρες χώρες. Από τη Συρία μέχρι τη Λιβύη είμαστε όλοι θύματα της τρομοκρατίας. Είμαστε θύματα μουσουλμά, μουσουλμάνοι, χριστιανοί, οι πάντες. Πρέπει να κινητοποιήσουμε κάθε πόρο που έχουμε για να αποκαταστήσουμε την σταθερότητα σε όλο τον κόσμο χρειάζεται να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις που έχουμε μπροστά μας και να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να χτυπήσουμε τους τρομοκράτες. Δεν πρέπει να απομονωθούμε, πρέπει να προσπαθήσουμε για να υπάρξει περισσότερη δημοκρατία. Του Κάτς για να έχουμε έναν από κάθε πολιτική ομάδα, ο κύριος Καστάλντο, για ένα λεπτό. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Οι πρόσφατες ε, τραγικές ε, τρομοκρατικές επιθέσεις σε διάφορες περιοχές του κόσμου πρέπει να μας οδηγήσουν να σκεφτούμε. Μιλάμε για τρομοκρατία σε κάθε ολομέλεια. Οι δρόμοι που μπορούμε να ακολουθήσουμε ωστόσο στην πράξη δύο παραμένουν. Πρώτον, αφενός να ακολουθήσουμε την, την αυταπάτη, να αποκλεινόμαστε, να βαφκαριζόμαστε ότι μπορεί να διασφαλίσουμε την ασφάλειά μας δαπανώντας περισσότερα σε όπλα, πληροφορίες, ασφάλεια. Σίγουρα θα είναι χρήσιμο κάτι τέτοιο, αλλά τελικά ε, θα μοιάζουμε με το παιδάκι που θέλει να βιάσει με ένα κοχύλι τη θάλασσα. Ή συνεχίζουμε να υποστηρίζουμε αυταρχικά καθεστώντας ελπίζοντας ότι το πρόβλημα θα λυθεί εκεί. Αυτό είναι ένα Λάθος που δεν το πληρώσουμε εν καιρό διότι δημιουργούνται άλλες συγκρούσεις. Αντίθετα μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε απευθείας ε, ζητώντας από το μετριοπαθές Ισλάμ στην Ευρώπη και στον Ισλαμικό κόσμο να γίνει ο μεγαλύτερος σύμμαχός μας, ο μόνος που μπορεί να απομονώσει την τρομοκρατία. Και τούτο μπορεί να γίνει αν μετέχει στην πολιτική ζωή. Πρέπει να επανεξετάσουμε λοιπόν την προσέγγιση μας για να βοηθήσουμε τις κυβερνήσεις αυτές να χτυπήσουν τις, ε, τους θύλακες φτώχειας, γιατί εκεί είναι η τρομοκρατία. Ευχαριστώ. Λόγο εκ μέρους της Επιτροπής έχει ο Επίτροπος κ. Δημήτρης Αβραμόπουλος. Κύριε Πρόεδρε, ο Parliament... Αξιότιμοι κύριοι βουλευτέ, καταρχήν σας ευχαριστώ όλους γιατί μου δίνετε σήμερα τη δυνατότητα να απαντήσω, να αντιδράσω και να σας παρουσιάσω την ανταπόκρισή μας στις απειλές που θέτουν οι τρομοκράτε. Δυστυχώς θα χρειαστεί πάρα πολύς χρόνος μέχρι να λυθεί το πρόβλημα αυτό και θα είμαι ευγνώμων διότι βάλατε το θέμα αυτό στην ημερήσια διάταξη αυτής της εβδομάδας συνόδου. Τους περασμένους έξι μήνες η Επιτροπή αυτή κατάφερε να προτείνει ορισμένα συγκεκριμένα μέτρα για να αντιμετωπίσει την απειλή αυτή. Πρέπει να συνεργαστούμε στις προσπάθειές μας για να βεβαιωθούμε ότι θα υπάρξει μία συνεχής και βιώσιμη εφαρμογή των προτάσεων αυτών σύμφωνα με, τα με σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων ταυτόχρονα. Σημείωσα αυτά που είπατε. Μερικοί ανέφεραν τα Δυτικά Βαλκάνια. Σας διαβεβαιώνω ότι και σε θέματα ασφαλείας τα Δυτικά Βαλκάνια είναι βασική μας εταίρη. Η σταθερότητα της περιοχής αυτής είναι ζωτική. εφαρμόζουμε στοχευμένες δράσεις στα Δυτικά Βαλκάνια κατά της ριζοσπαστικοποίησης και συνεργασία για την καταπολέμηση λαθρεμπορίας όπλων. Πολλοί από εσά τόνισαν όπως είναι φυσικό το θέμα της τυνησίας. Κατά την εισήγησή μου, την αρχική μου εισήγηση, και εγώ αναφέρθηκα στην Τινησία που είναι εταίρος μας και τον υποστηρίζουμε πλήρως, την υποστηρίζουμε πλήρως στα πλαίσια της αναθεώρησης της ευρωπαϊκής πολιτικής γειτονίας θα αναπτύξουμε κι άλλες στοχευμένες δράσεις για την Τινησία. Τις επεξεργαζόμαστε αυτή τη στιγμή μαζί με την κυρία Μογκερίνη και τον Επίτροπο Χάν. Και ήδη αρχίσαμε να έχουμε αποτελέσματα. Είμαι σίγουρος ότι στις ε, προσεχείς συζητήσεις θα το ξαναπούμε αυτό. Αλλά σας επαναλαμβάνω ότι είμαι δεσμευμένος να συνεργαστώ χέρι με χέρι με το Κοινοβούλιο και φυσικά το Συμβούλιο για αυτό το θέμα. Υπολογίζω πραγματικά στην υποστήριξή σας. Σας ευχαριστώ. Το λόγο έχει εκ μέρους του Συμβουλίου ο Σμιτ. Monsieur le Président, euh, euh, Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι βουλευτές, όλοι συμφωνούμε ότι είναι κατεπήγον το θέμα. Πρέπει να εντατικοποιηθεί η συνεργασία μας σε διάφορους τομείς και να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα τόσο δίωξης όσο και πρόληψης. Πρέπει επίσης να υπάρξει μια συστηματική προσέγγιση και ολοκληρωμένη αλλά χωρίς να μπούμε να πέσουμε στο λάθος της ξενόη Ισλαμοφοβίας και του στιγματισμού γιατί τότε παίζουμε το παιχνίδι των τρομοκρατών. Πρέπει να συνεχίσουμε να στηρίζουμε τις τρίτες χώρες με τις οποίες έχουμε δεσμευθεί να συνεργαστούμε για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας μέσω συνδυασμένων προγραμμάτων και όπως είπε και ο Επίτροπος προβλέπεται ήδη η συζήτηση για την πολιτική γειτονία σαν μόλις ήρθε και ο Επίτροπος Αν και για χώρες όπως η Τινησία που είναι ιδιαίτερα ευάλωτες και που πρέπει να τις στηρίξουμε ενεργά. Η μονάδα που ασχολείται για το περιεχόμενο των διαφόρων αναρτήσεων στο Ιντερνετ επίσης είναι κάτι πολύ χρήσιμο και πρέπει να το προωθήσουμε. Και επιτρέψτε μου επίσης να πω καταλήγοντας ότι θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να υπάρξει συμφωνία για την οδηγία PNR της Ευρώπης κατά την Προεδρία μας. Να ξέρετε ότι η Προεδρία θέλει να επεξεργαστεί αυτό το θέμα αποτελεσματικά σε στενή συνεργασία με το Κοινοβούλιο σας, επί του οποίου υπολογίζουμε. Ευχαριστώ. Το επόμενο θέμα στην ημερήσια διάταξη είναι δήλωση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής ΥΠΑΤΗ είπα εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας